Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να συνεχίσουμε τώρα με το σημείο 9 της ημερήσιας διάταξης, αλλά δεν είναι εδώ ακόμη ο εισηγητής. Αν μου επιτρέπετε, να πάμε στο σημείο 11. Καταρχάς γιατί εγώ είμαι ο εισηγητής για το θέμα αυτό άρα είναι ευκολότερο. Το σημείο 11 αφορά ενημέρωση της Επιτροπής σε σχέση με την οδηγία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων. Εχθές στις 20 ε, Φεβρουαρίου έγινε ο πρώτος τριμερής διάλογος ε, για την πρόταση κανονισμού σε σχέση με τους κανόνες για την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων που είναι ο πλήρης τίτλος ε, του κανονισμού. Ε, η διαπραγματευτική εντολή του Κοινοβουλίου εγκρίθηκε στην Επιτροπή μας τον Νοέμβριο του 2017 και ε, επιβεβαιώθηκε από το Κοινοβούλιο βάσει του κανόνα 69 συν του εσωτερικού κανονισμού. Ο εισηγητής για το θέμα αυτό ε, αποχώρησε και είναι σκιώδης εισηγητής για την ομάδα των σοσιαλιστών και δημοκρατών. Οπότε έχω αναλάβει εγώ την ευθύνη για το θέμα αυτό. Ο κύριος στόχος αυτού του πρώτου τριμερούς διαλόγου ήταν ε, να παρουσιάσουν και να εξηγήσουν τις θέσεις των ε, ε, αντίστοιχων οργάνων ε, για το θέμα αυτό και να συνεχίσουν σε μια εντολή για την συνέχεια της δουλειάς, μεταξύ το, της οποίας βέβαια υπάρχει και προπαρασκευαστική δουλειά σε τεχνικό επίπεδο. Το, η διαπραγματευτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχε μια επικοδομητική ε, ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο Γκάμπριελ και την ε, πρέσβη Γκάμπ, Κόνεβα ε, και συζήτησαν ειδικότερα το θέμα της επέκτασης του πεδίου εφαρμογή της αρχής προέλευσης, ε, τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων, την ε, ε, τεχνική direct injection και γενικότερα το πεδίο εφαρμογή του κανονισμού. Ο δεύτερος και ο τρίτος τριμερής διάλογος θα λάβει χώρα στις συνόδους του Στρασβούργου το Μάρτιο και τον Απρίλιο. Αυτά έχω να σας πω εγώ. Θέλει κανένα συνάδελφος να σχολιάσει αυτή την ενημέρωση? Μάλλον όχι. Και επειδή ήρθε τώρα και ο κύριος Μαστάλκα, μπορούμε να συνεχίσουμε με το σημείο 9, που είναι η εξέταση των τροπολογιών για το καταστατικό επιχειρήσεων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Κύριε Μαστάλκα, έχετε το λόγο. Συγγνώμη που άργησα. Νομίζω ότι πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των παράλληλων συνεδριάσεων ή τα χιλιόμετρα των διαδρόμων και διαδρομών που έχουμε να κάνουμε. Για να φτάσουμε εδώ δεν αντέχει η καρδιά μου. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω όλους ε, τους συναδέλφους για τις τροπολογίες ε, που υπέβαλαν στην έκθεσή μου για το καταστατικό επιχειρήσεων κοινωνικής και αλληλέγγυα οικονομίας. 165 τροπολογίες λάβαμε συνολικά που αφορούν κυρίως τους εξής τομείς. Πρώτον, τον ορισμό κοινωνική οικονομία και επιχείρηση κοινωνικής οικονομίας. Δεύτερον, δίνεται έμφαση στον σημαντικό ρόλο που παίζει η κοινωνική οικονομία στην οικονομία εν γέννη. Τρίτον, υπογραμμίζουμε πως οι νόμοι και οι κανονισμοί στα κράτη-μέλη ποικίλουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Γι' αυτό και επηρεάζεται και το τι ακριβώς ε, χαρακτηριστικά έχουν επιχειρήσει κοινωνικής και αλληλεγγύης οικονομίας σε κάθε χώρα. Έπειτα, η διαχείριση αυτών των επιχειρήσεων, η... το σήμα, το επόμενο, το κοινωνικό σήμα και το επόμενο κριτήρια για να πάρει κανείς αυτό το σήμα. Περισσότερε τροπολογίες νομίζω ότι μπορούν να, ε, να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο των συμβαστικών τροπολογιών. Αυτό που δημιουργεί πρόβλημα όμως είναι κυρίως τροπολογίες σε 39 έως 43 και 45 έως 47 τροπολογίες από συναδέλφους της ομάδας ΙΕΝΕΦ. Στόχος τους είναι να απαλληφθούν σημαντικά στοιχεία των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας. Έχουμε και την τροπολογία 96 και τις επόμενες, οι οποίες διαγράφουν την ιδέα περί Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Σήματος, European Social Label. Καταλαβαίνω ότι οι συνάδελφοι από το ΙΕΝΕΦ είναι εναντίον ουσδήποτε εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ωστόσο, θέλω να τους πω το εξής. Οι εκπρόσωποι των ίδιων αυτών των επιχειρήσεων ζήτησαν να υπάρξει μια αναρμονισμένη προσέγγιση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή αυτό που κάνουμε είναι ε, μια προσπάθεια να διευκολύνουμε την πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις στις εταιρείε αυτές, που θα είναι πιο εύκολα να γνωρίσουμε χάρη σε αυτό το σήμα. Θα μπορούσαμε ίσως οι συνάδελφοι από το ΙΕΝΕΦ να μας εξηγήσουν τι θέλουν να πετύχουν τις τροπολογίες τους. Κυρία Ρέγκνερ, δεν τη βλέπω βέβαια εδώ, ε, και αυτή θα ήθελα να μου εξηγήσει την τροπολογία της. Αλλιώς βέβαια μπορούμε να το συζητήσουμε διμέρως αν δεν έρθει. Δεν νομίζω ότι έχουμε μεγάλες διαφορές με τους σκιώδες ό,τι αφορά τη γενική κατεύθυνση και προσανατολισμό της έκθεσης πλήν των τροπολογιών ENF. και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να αρχίσουμε ήδη να δουλεύουμε πάνω στις συμβαστικέ προτάσεις. Ε, έχουμε τις τροπολογίες ε, γραπτός, έχουμε και χρόνο γιατί ζητήθηκε και μια μικρή αναβολή στο χρονοδιάγραμμα και θα ψηφίσουμε επομένως το Μάιο στην Επιτροπή. Ευχαριστώ για την προσοχή και προσβλέπω στη συνεργασία με όλους τους συναδέλφους. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος ε, Ραϊεφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα για μια ακόμη φορά να συγχαρώ τον κύριο Μαστάλκα για την πολύ καλή και ισορροπημένη έκθεση που έχουμε αναχείρας. Έχουν κατατεθεί πράγματι πολλές τροπολογίες και είμαι βέβαιος ότι πολλές εξ αυτών θα συμβάλλουν στο να είναι πολύ καλύτερη η τελική εκδοχή του κειμένου. Μελέτησα τις τροπολογίες και μπορώ να πω ότι μου κίνησαν την προσοχή κάποια σημεία. Το πρώτο, και πρέπει να το τονίσουμε, είναι ότι στόχος της πρότασης αυτής είναι ένα που πρέπει να επιτευχθεί εντό των αρμοδιοτήτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα θα πρέπει να γίνουν σεβαστέ οι αρχέ τη αναλογικότητα και τη επικουρικότητα. Χωρί τα κράτη-μέλη να απαιτηθεί να προβούν σε μείζονε αλλαγέ ε, του εταιρικού δικαίου ή των ρυθμιστικών του συστημάτων. Δεύτερον, και θεωρώ ότι είναι και σημαντικό αυτό, θα πρέπει να μελετήσουμε πολύ προσεκτικά το ζήτημα της χαμηλής κερδοφορίας αυτών των επιχειρήσεων. Κάποιοι συνάδελφοι έφτασαν στα άκρα. Δηλαδή ε, απορρίπτουν τον οποιοδήποτε είναι κερδοφορίας για αυτές τις επιχειρήσεις. Δεν πιστεύω όμως ότι πρέπει να κατηγορούνται αυτές οι επιχειρήσεις αν κερδίσουν ε, χρήματα. Απλά το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους θα πρέπει να φροντίσουμε να επανεπενδύεται σε αυτές τις επιχειρήσεις και στις ε, δραστηριότητές τους γιατί έχουν ένα πρωταρχικό στόχο που πρέπει να υπηρετούν και αυτόν τον στόχο εκεί θα πρέπει να πηγαίνουν αυτά τα χρήματα. Δηλαδή κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Και τέλος, υπάρχουν ενδιαφέρουσες προτάσεις που αφορούν ασφαλιστικές δικλείδες, εχέγγυα αλλά και κυρώσεις αν υπάρξει κατάχρηση του κοινωνικού αυτού επιχειρηματικού σήματος. Αν θέλουμε να καταστεί επιχειρησιακό αυτό το σύστημα θα πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρά όλες οι αρχές για αυτό το σήμα και θα πρέπει οι αγορές να αναγνωρίζουν το σήμα για να μην, να μην υπάρχει διακριτική μεταχείριση των εταιριών ανάλογα με το κράτος μέλους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αντελβό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη εξ ονόματος της κυρίας Ροζιέρ που είναι σκιώδης και θα σας διαβάσω τις σκέψεις της και ζητώ συγγνώμη ε, από τον κύριο ε, Μαστάλκα γιατί δεν μπορώ να δώσω εγώ την απάντηση από τη συνάδελφο. Καλωσορίζω τις ενδιαφέρουσες προτάσεις μέσω τροπολογιών για να ε, ευοδοθεί αυτό το σχέδιο. Έχει υποβάλει τροπολογίες υπ' αυτή την έννοια, εκ των οποίων απορρέουν οι εξής ιδέες. Δεν πρέπει να μειώσουμε το εύρος των επιχειρήσεων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή την ονομασία και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι δρούν μόνο στο κοινωνικό τομέα, αλλά είναι, λειτουργούν σαν επιχειρήσεις κοινή ωφελία έτσι ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των πολιτών καθώς και ε, η φυσική και πολιτιστική κατάστασή τους. Το πεδίο εφαρμογής επίσης δεν θα πρέπει να περιοριστεί στις επιχειρήσεις δουν ως μη κερδοσκοπικές. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε το ρόλο των κερδοσκοπιών, κερδοσκοπικών επιχειρήσεων καθώς και τις επιχειρήσεις με περιορισμένο κερδοσκοπικό χαρακτήρα μέσα στα πλαίσια των απότερων στόχων τους. Αυτές οι επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να θεωρηθούν κερδοσκοπικού χαρακτήρα και θα πρέπει να ε, μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τα μέτρα αυτά. Επίσης, ε, δεν θα πρέπει να υπάρχει συσταλτική ερμηνεία αυτών των επιχειρήσεων. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα κριτήρια δημοκρατικής διακυβέρνησης που θα πρέπει να προσέξουμε, διότι σχετίζονται με την αλληλέγγυα οικονομία και με την ίση συμμετοχή όλων. Και ως προς τη διαφορά των μισθολογίων θα μπορούσαν να φυγούν από αυτή την έκθεση. Ορισμένες προτάσεις προτείνουν να δοθεί η ευκαιρία στα κράτη-μέλη ε, να αποδώσουν αυτό τον τίτλο στις επιχειρήσεις ε, η κυρία Ροζιέρ θεωρεί ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε για εναρμονισμένη προσέγγιση, ακόμα και αν αυτό είναι ο απότερος στόχος ε, της έκθεσης. Η έκθεση αυτή θα πρέπει να ορίσει κοινά κριτήρια για να μπορέσουμε να έχουμε ένα συνεκτικό πλαίσιο κοινωνικού μελήματος και αλληλεγγύης. Άρα ε, μας απασχολεί το γεγονός ότι πολλοί συνάδελφοι καθιστούν το γράμμα της πρότασης κενό περιεχομένου. Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία έχει μεγάλη σημασία για την εσωτερική αγορά μέσα στα πλαίσια της καινοτομίας, της ανθεκτικότητας και της δυνατότητας ε, καταπολέμησης της ανεργίας και του αποκλεισμού. Η κυρία Ροζιέρ θέλει να συνεργαστεί με τον εισηγητή και με τους άλλους ε, συναδέλφους, τους οποίους ευχαριστεί εκ των προτέρων. Σας ευχαριστώ. Δεν ε, ζητά κανένας άλλος το λόγο. Α, ναι, με συγχωρείτε. Ο κύριος Ντυρά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι σκιώδης επί του θέματος και μια και είμαι και παρόν, θα ήθελα να λάβω το λόγο. Καταρχήν για να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εργασία του, να του πω ότι θα τον υποστηρίξουν πλήρως οι πράσινοι σε, αυτό το, σε αυτή την έκθεση για να δημιουργήσουμε μία νέα ορατότητα στην οικονομία αυτή που αφορά 14 εκατομμύρια πολίτες και θέλουμε να υποστηρίξουμε πλήρως την έκθεσή σας περί κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, έτσι ώστε να έχει σαφή αντίκτυπο. Δεν μπορώ να απαντήσω για την κυρία ε, ε, Ρέγνερ και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν, ε, γίνονται ορισμένες διαγραφές που θα προωθούσαν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Les entrepreneurs européens, il est de faire en sorte que l'Europe και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλοί θέλουν να εξαφανιστεί η Ευρώπη από το χάρτη ιδιαίτερα από πλευράς ε, Ευρώπης των Εθνών. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να αποκαταστήσουμε τα πράγματα. Λυπάμαι για τους απόντες. Επί της ουσίας, οι δικές μας τροπολογίες αφορούν ένα βασικό σημείο στη Γαλλία και όχι μόνο στη Γαλλία, τον τομέα της υγείας. Όπως ξέρετε, οι υπηρεσίες υγείας εντάσσονται στις επιχειρήσεις κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Θα πρέπει να ενισχυθούν αυτές οι επιχειρήσεις, όπως είπε και η κυρία Ροζιέρ, το, με το θέμα το, της διακυβέρνησης και συμμερίζουμε την άποψη της κυρίας, της κυρίας Ροζιέρ γιατί υπάρχουν κερδοσκοπικά στοιχεία και χαρακτήρας που θα πρέπει να μας απασχολήσουν είτε στα κέρδη είτε οπουδήποτε αλλού για αυτές τις επιχειρήσεις ε, ε, κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Και τίθεται και ένα άλλο ζήτημα των ενδεχομένων κυρώσεων τη στιγμή που δεν λαμβάνεται υπόψη αυτή η διατύπωση και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αν χάσει κανείς αυτό τον ε, τίτλο θα πρέπει να δούμε σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Ποιο θα είναι το, το νομικό καθεστώς που θα διέπει αυτές τις επιχειρήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ για τον συνενετικό τρόπο που θίξατε αυτά τα ζητήματα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ίσως ο κύριος Μαστάλκα θέλει κάτι να προσθέσει. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για όλα τα στοιχεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία σας. Ο κύριος Ραντέφ και εγώ συζητήσαμε ορισμένα από τα ζητήματα που εφήγησαν και εδώ. Νομίζω ε, ότι δεν μιλάμε για τον κερδοσκοπικό χαρακτήρα που είναι η βάση, γιατί μπορεί να υπάρχουν κέρδη, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να συμβαδίζουμε με μια ορθολογική σκέψη σε σχέση με τον τρόπο δηλαδή διατύπωσης θα πρέπει να ορίσουμε ένα πλαίσιο διατύπωσης και να δούμε και τις ενδεχόμενες κυρώσεις που θα είχαν επίπτωση. Θα φτάσουμε στη συνένεση εκτός από συναδέλφους από μία πολιτική ομάδα, αυτή είναι η δημοκρατία, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, αλλά φαίνεται ότι κινούμαστε προς την σωστή κατεύθυνση, όπως λένε οι συνάδελφοι. Θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μήπως να λάβει το λόγο, συγγνώμη σας ξέχασα. Μάλλον όχι. Οπότε να ολοκληρώσω αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης λέγοντας ότι η έγκριση στην Επιτροπή μας έχει προγραμματιστεί για τη συνεδρίασή μας ε, στις 14 και 15 Μαΐου του 2018. Να συνεχίσουμε τώρα με το σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης που είναι η εξέταση του σχεδίου έκθεσης για την παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2016 Δίνω το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Χρυσόγονο. Thank you, Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, η σωστή εφαρμογή της, ε, του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι βασικό στοιχείο για την ε, βελτίωσή της. Σε αυτό το πλαίσιο, η προσεκτική και αντικειμενική παρακολούθηση των κρατών μελών ε, και των δράσεων και παραλήψεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ μεγάλη σημασία. Η εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη σωστή και έγκαιρη μεταγραφή της ε, ενωσιακής νομοθεσίας, γιατί διαφορετικά στερούνται οι επιχειρήσεις και οι πολίτες από τα ωφέλη που απορρέουν. Γι' αυτό η, η έκθεση για την παρακολούθηση της εφαρμογής ε, του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα περιορίζεται μόνο σε μία μεμονωμένη παρουσίαση επισήμων στοιχείων. Ναι. Αντιθέτως, ε, δείχνει τις αδυναμίες της εφαρμογής ε, του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο αντίκτυπος αυτών ε, των μείων εκτιμάτων της ανεπαρκούς εφαρμογής θα διερευνηθούν επαρκώς και θα προταθούν ρεαλιστικές λύσεις. Σε γενικέ γραμμέ, η έκθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρακολούθηση τη εφαρμογή του δικαίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση το 2016 φαίνεται να μην λαμβάνει υπόψη ε, πλήρω αυτού του στόχου. Ε, η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2016 και την εφαρμογή της ενωσιακής, του ενωσιακού δικαίου αναφέρει ότι οι, χώρες, ε, ότι οι περισσότερες επιπαραβάσει διαδικασίες αφορούσαν το, η δικαιοσύνη, και του καταναλωτέ το περιβάλλον, τη φορολόγηση και την εσωτερική αγορά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε 3.783 καταγγελίες που ανέφεραν ενδεχόμενη παραβίαση της ενωσιακής νομοθεσίας με την Ιταλία, την Ισπανία και τη Γαλλία που είναι, να είναι τα κράτη-μέλη κατά των οποίων ε, ε υπευλήθησαν οι περισσότερες καταγγελίες. Ε, πρέπει να τονίσουμε ότι ο αριθμός των καταγγελιών ε, είναι ε, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2011. Το υψηλό επίπεδο επιπαραβάσει διαδικασιών το, το 2016 έφτασε σε μία περίοδο εχμής 5 ετών και αυτό δημιουργεί μεγάλες ανησυχίες. Από την άλλη, η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φαίνεται να παραγνωρίζει ότι τα προγράμματα προσαρμογής που εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη και που προωθούνται από τους θεσμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν επηρεάσει σοβαρά τα θεμελιώδη δικαιώματα μεταξύ των οποίων την πρόσβαση στη στέγαση, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την εκπαίδευση, τη δικαστική προστασία και τα εργασιακά δικαιώματα. Επειδή όλοι οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεσμεύονται από τις συνθήκες της Ένωσης και από τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης, το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ Ευρωπαϊκών Οργάνων και ε, κρατών μελών πρέπει να θεωρούνται, κατά τη γνώμη μου, ε, πράξεις ε, δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φαίνεται όμως αυτό να αντιβαίνει στις θεμελιώδεις αρχής Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι τα καθήκοντα που εχωρούνται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στην Επιτροπή στο πλαίσιο της συνθήκης δεν σημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα να λάβουν απόφαση από μόνοι τους. Οι δραστηριότητες αυτών των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός της συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης δεσμεύουν μόνο τον ESM και όχι ε, τα, ε, ε, τους θεσμούς της Ένωσης. Ε, οι βασικές, οι κύριες αποφάσεις, οι σημαντικότερες αποφάσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τους πολίτες και για τα κράτη-μέλη, όπως οι αποφάσεις για τους εθνικαίους προπολογισμούς και τις μεταρρυθμίσεις, λαμβάνονται από τους Υπουργούς Οικονομικών ε, στο Eurogroup, χωρίς επίσημους κανόνες και χωρίς πολλή διαφάνεια. Και το αποτέλεσμα είναι ότι δεν υπάρχει αρκετή λογοδοσία ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα άλλα θεσμικά όργανα. Πέρα από αυτό όμως πρέπει να τονιστεί ότι οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη-μέλη θα δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή των μέτρων που εγκρίθηκαν στον τομέα ε, του ασύλου και της μετανάστευσης ώστε να εξασφαλιστεί ότι συμμορφώνονται πλήρως με τις αρχές ε, που συμπεριλαμβάνει η Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη-μέλη θα ανταποκριθούν αποτελεσματικά στην ε, εξελισσόμενη κατάσταση ασφάλειας και μετανάστευσης, ε, θα επιβάλλουν το θεματολόγιο το σχετικό με τη μετανάστευση, όπως επίσης και τα σχετικά πακέτα εφαρμογής. Οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ενθαρρυνθούν ε, να αναλάβουν σε κάθε χρονική στιγμή το καθήκον τους του σεβασμού ε, του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το παράγωγο δίκαιο ε, και αυτό θα ε, συμβαίνει επίσης και όταν ε, λαμβάνονται αποφάσεις για πολιτικές ή συνάπτουν συμφωνίες με φορείς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης θα ενθαρρύνονται να αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους, να επικουρούν τα κράτη-μέλη με κάθε διαθέσιμο μέσος προς τη μεταγραφή της ενωσιακής νομοθεσίας σε όλους τους τομείς, δείχνοντας συνεργασία και αλληλεγγύη στους πιο αδύναμους εταίρους. Και όπως ε, είχε πει και ο Αριστοτέλης ε, πριν από 24 αιώνες, ο νόμος θα υπηρετεί την κοινωνία και δεν θα είναι ένας τύρανος που θα κάνει την κοινωνία και τους πολίτες να υποφέρουν. Αντιθέτως, η εφαρμογή ε, του νόμου θα οδηγήσει σε μια αηφόρο ευημερία της κοινωνίας και τους πολίτες τους. Ευχαριστώ. Um, Θέλει κάποιος το λόγο, κυρία Ντελβό. Αυτή τη φορά εκπροσωπώ την κυρία Κάφμαν. Η κυρία Κάφμαν ευχαριστεί τον εισηγητή, τον κύριο Χρυσόγωνο, για το σχέδιο έκθεσής του. Πολύ σύντομα θα ήθελα να τονίσω δύο στοιχεία τα οποία η κυρία Κάφμαν θεωρεί σημαντικά. Ε, το υψηλό ποσοστό ε, των διαδικασιών επί παραβάση το 2016 δείχνουν ε, ότι στα κράτη-μέλη η εφαρμογή των κανόνων από τα κράτη-μέλη εξακολουθεί να παραμένει μεγάλη πρόκληση που συνοδεύεται από σημαντικές απαιτήσεις. Το 2016 σε ό,τι αφορά τις ε, νέες καταγγελίες ε, είχαμε το μεγαλύτερο αριθμό ρεκόρ μετά το 2011. Αυτό είναι σημαντικό και έχει να κάνει και με τις ε, καταναλωτικές διαφορές η αύξηση αυτού του ποσοστού. Και όλα αυτά που καταδεικνύουν ότι μπορεί να υπάρξει περιορισμός των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των καταναλωτών στα κράτη-μέλη πρέπει όμως να εφαρμόζονται οι διατάξεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Χρειάζεται καλή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι σημαντικό ιδίως για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου. Επίσης είναι σημαντικός και ο μεγάλος ρόλος των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών για την εξεργασία των κανόνων και για να μην υπάρχουν καθυστερήσεις και ε, παραλήψεις από τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν ε, κάνει τίποτα λέει ο Πρόεδρος. Μέχρι πού φτάνει αυτή η αντιπροσωπευτική δημοκρατία, διαρωτώ με. Κυρία Χάουταλα. I, I just come from Μόλι βγήκα από μια συνάντηση με την κοινότητα των πολιτών, όπου τουλάχιστον 11 ευρωβουλευτέ διαφορετικών επιτροπών και διαφορετικών πολιτικών ομάδων ήταν παρόντε. Και ο κ. Χερμπράντι είπε στο κοινοβούλιο, όταν συνεδριάζουν κοινοβουλευτικέ επιτροπέ, δεν έχουμε ξαναδεί τόσου πολλέ βουλευτέ στην αίθουσα. Τέλο πάντων, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Χρυσόγονο για την δουλειά του, πολύ διεξοδική και αυτή τη φορά σε ό,τι αφορά την ε, παρακολούθηση της εφαρμογής ε, του δικαίου το 2016. Πολλές φορές ε, ο ένας αντικαθιστά τον άλλον από τον ένα στον άλλο. Το θέμα είναι ότι σίγουρα απαιτείται νομική εξέταση του ζητήματος και δει πόσο η ΕΚΤΑ, ο μηχανισμός σταθερότητας του ESM δηλαδή, μπορούν να υπαγορεύουν μέτρα που δημιουργούν για ένα κράτος μέλος και τους πολίτες του μια κατάσταση που ουσιαστικά παραβιάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα. Αυτό δεν πρέπει να το δούμε ακροφυγός ούτε ελαφρά. Και ήταν και μια έκθεση, ήταν μάλλον ε, και μια παρατήρηση στην έκθεση του κυρίου Χρυσόγνου πριν από δύο-τρία χρόνια. Πρέπει να το δούμε σοβαρά λοιπόν. Επίσης, νομίζω ότι είναι χρήσιμο που ζητείτε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή μέτρων στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης. γιατί πρέπει να είναι τελείως διαφορετική αντιμετώπιση ανάλογα με το κράτος μέλος από ό,τι φαίνεται. Ενώ πρέπει να τηρούνται αρχές του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Άρα θα μπορούσαμε να εμβαθύνουμε. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή σε πολλά κράτη-μέλη γίνεται μια συζήτηση για την επιστροφή έτου τον άσυλο που δεν τους χορηγείται άσυλο, γιατί δεν ε, τους αναγνωρίζεται το καθεστώς του πρόσφυγα. Και γίνεται η συζήτηση για το πώς εφαρμόζεται το σύστημα από άλλα κράτη-μέλη. Μπορούμε λοιπόν και εμείς να εμβαθύνουμε σε αυτό. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Αν δεν υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι, θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει το λόγο. Όχι. They might have their reasons. Θα έχουν τους λόγους τους. Οπότε, το μόνο που έχω να προσθέσω είναι ότι η προθεσμία κατάθεσης ε, τροπολογιών είναι η 28 η Φεβρουαρίου, 12 το μεσημέρι. Και τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε το σημείο 10, που είναι η ενημέρωση της Επιτροπής ε, για το θέμα των συμβάσεων για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου. Έχουμε εδώ την κυρία Γκέπχαρτ. Είναι η μία από τους δύο συνεισηγητές. Λείπει ο κύριος Φως. Οπότε, κυρία Γκέπχαρτ, έχετε εσείς το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σας ευχαριστήσω που μας δίνετε τη δυνατότητα να σας ενημερώσουμε για το πώς, προχωρούν οι συνομιλίες στο πλαίσιο του τριμερούς διαλόγου για το ψηφιακό περιεχόμενο. Πρέπει να σας πω ότι και από πολιτικής και τεχνικής πλευράς και με την προηγούμενη και με την Προεδρία του Συμβουλίου έχουμε συνεργαστεί πολύ ε, καλά και έχουμε καταφέρει να βρούμε καλές λύσεις. Και νομίζω ότι είναι και αυτό μια πολύ σημαντική προϋπόθεση αν θέλουμε να σημειώσουμε πρόοδο. Ένα που μπορώ να πω πολύ ξεκάθαρα εδώ είναι ότι όπως εξελίσσονται αυτές οι συνομιλίες μπορώ να φανταστώ ότι επί βουλγαρικής προεδρίας θα μπορούσαμε να καταλήξουμε να έχουμε δηλαδή ένα θετικό αποτέλεσμα αυτού του τριμερούς διαλόγου. Και αυτό είναι πολύ θετικό, διότι ακριβώς στον τομέα αυτό είναι σημαντική η πρόοδος, πρέπει να επιτευχθεί πρόοδος. Επομένως, ήδη έχουμε συμφωνήσει σε πολλά σημεία δεν έχω πολύ χρόνο για να αναφέρω δεξιοδικά όλα αυτούς τους τομείς γιατί είναι πάρα πολλοί. Τρεις τομείς ακόμα χρήζουν περαιτέρω ε, συνεννόησης ε, και συζητήσεων μεταξύ των τρινοθεσμικών οργάνων. Το ένα θέμα αφορά ε, το βαθμό εναρμόνισης σε ό,τι αφορά τις προθεσμίες για την παροχή των ψηφιακών υπηρεσιών. Το Συμβούλιο θέλει την ελάχιστη δυνατή εναρμόνιση. Εμείς βέβαια ως Κοινοβούλιο ξεκαθαρίσουμε ότι ε, χρειαζόμαστε ως το δυνατόν πληρέστερη εναρμόνιση. Είμαστε εδώ σε έναν τομέα που και στη Βρετανία και στην Ολλανδία δεν υπάρχουν ε, σχετικές διατάξεις ε, και γι' αυτό είναι σημαντικό να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες όλα τα κρατημέλη. Αυτό είναι ένα σημείο που πρέπει ακόμη να επεξεργαστούμε. Ένα δεύτερο σημείο όπου έχουμε προβλήματα είναι ο κανονισμός ε, για τα, δικαιώματα προσωπι... για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ε, και το... στις παραβιάσεις αυτού του κανονισμού. Γνωρίζετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ξεκαθαρίσει ότι εμείς ε, ε, είμαστε κατά ε, του data mining σε ό,τι αφορά την ε, συμμόρφωση προς την οδηγία για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Δεν το θέλει το Συμβούλιο. Εμείς έχουμε αποφασίσει να διοργανώσουμε μία νέα ακρόαση με τους εμπειρογνώμονες. Έγινε, καλέσαμε Κομισιόν και Συμβούλιο και τι είχαμε τελικά, έναν εμπειρογνώμονα υπέρ, έναν κατά και το αποτέλεσμα αυτών των ε, ακροάσεων ήταν ότι και οι δύο εμπειρογνώμονε στήριξαν την υπόθεση ότι ε, θα υπάρχει ασφάλεια δικαίου αν υπάρχει ε, τουλάχιστον μία αρχή στην μία περίπτωση παραβίασης της οδηγίας των για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Το θέμα είναι ότι θέλουμε να έχουμε ε, πραγματικά σαφήνεια και ασφάλεια δικαίου και να μην ε, παρακάμψουμε το πρόβλημα. Ελπίζω να το καταφέρουμε και να πείσουμε και το Συμβούλιο. Το περίεργο είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε κάνει τη σχετική πρόταση και κατά το παρελθόν, αλλά το Συμβούλιο δεν μας διευκολύνει. Νομίζω όμως ότι είναι πολύ σημαντικό για την προστασία των καταναλωτών. Το είπαν και ξεκάθαρα οι δύο εμπειρογνώμονες, οπότε ελπίζω να πείσουμε και τα κράτη-μέλη. Αυτό θα το προσπαθήσουμε τουλάχιστον. Το τρίτο σημείο που υπάρχει ακόμη απόκληση απόψεων είναι τα ενσώματα μέσα, δηλαδή τα προϊόντα που έχουν ενσωματωμένα ψηφιακά περιεχόμενα, ψηφιακέ υπηρεσίε, ηλεκτρονικό αυτοκίνητο, iPad κτλ. Με τον ε, εισηγητή ε, Αριμό και την κυρία Χάουταλα ε, είχαμε το άρθρο 450 και έχουμε προσπαθήσει να διευκρινίσουμε ξεκάθαρα ότι εντάσσεται στην οδηγία για το ψηφικό περιεχόμενο το σύνολο των ψηφιακών ε, προϊόντων και υπηρεσιών. Θα ήταν περίεργο να έχουμε διαφορετικά ε, νομοθετήματα να ισχύουν και διαφορετικά δικαιώματα να κατοχυρώνονται όταν έχουμε μια προκατεστημένη εφαρμογή στο κινητό μας τηλέφωνο ε, και να ισχύει ένα συγκεκριμένο ε, σετ κανόνων. Όταν εγκαθαστήσουμε μια νέα εφαρμογή, να η επικαιροποιήσουμε την εφαρμογή αυτή, να αλλάζει οι κανόνες που εφαρμόζονται. Και εμείς έχουμε πει ότι θα πρέπει να υπάρχει μια διατήρηση ε, των κανόνων, γιατί τέλος αυτό δημιουργεί προβλήματα στους καταναλωτές, πολιτές, ε, στους ε, κατασκευαστές και δεν υπάρχει ασφάλεια δικαίου. Δεν ε, καταλαβαίνω ακριβώς γιατί το Συμβούλιο είναι κατά. Από ό,τι δεν άκουσα, το Συμβούλιο συζητά μια νέα παραλλαγή για το άρθρο 20 της οδηγίας. Δεν ξέρω πώς λέγεται αυτή η οδηγία για αυτά τα ε, αγαθά Αν γίνει αυτό δεν θα προσπαθήσω να το αποδίσω, Θέλω να το συζητήσω βέβαια και με τον ε, εισηγητή Φώσο γιατί δεν το έχω ακόμη καταφέρει. Αλλά αν πραγματικά αυτό μας δώσει μια λύση νομίζω ότι είναι κάτι θετικό. Οπότε μπορούμε να δείξουμε ευελιξία. Αυτά είναι τα τρία σημεία λοιπόν για τα οποία απαιτούνται περαιτέρω συζητήσεις, αλλά οι συζητήσεις με την Προεδρία του Συμβουλίου είναι χαρακτηρίζονται από πνεύμα συνένεσης. Δεν υπάρχουν δηλαδή ε, αν μπορώ να το πω έτσι, ε, περιχαρακωμένες απόψεις και νομίζω ότι μέσα στο επόμενο τρίμηνο θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε μια ε, απόφαση. Τα τεχνικά, οι τεχνικές συναντήσεις πηγαίνουν πολύ καλά και ο τριμερής διάλογος επόμενος προβλέπει προβλέψεις 16 Μαρτίου. Εκεί θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον από τα τρία σημεία αυτά να το αποκρισταλώσουμε και νομίζω τότε θα είμαστε και σε καλό δρόμο. Ευχαριστώ. Any observations from the... Παρατηρήσεις υπάρχουν από τους συναδέλφους κυρία Χάουταλ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, συμφωνώ με την κυρία Γκέπχαρτ. Όποια δηλαδή και να είναι η απόφαση για το ενσωματωμένο ψηφιακό περιεχόμενο, για τα ενσώματα αγαθά ή όχι, θα πρέπει να δούμε πώς θα έχει η όλη εξέλιξη του ζητήματος γενικότερα. Τι πιστεύετε σε σχέση με τα ε, ενσώματα αγαθά διότι όπως ξέρετε δεν υπήρξε ε, πλειοψηφία για ε, μέγιστη εναρμόνιση ούτε για ελάχιστη. Αυτό ε, θα προδικάσει τα ζητήματα που θα ανακύψουν όταν τα κράτη-μέλη αρχίσουν να συζητούν αυτό το ζήτημα. Τι πιστεύετε ότι θα συμβεί με την ψήφιση αυτή της έκθεσης. Νομίζω ότι αύριο θα ψηφιστεί η έκθεση στην ΙΜΚΟ. Ναι, πράγματι αύριο θα ψηφιστεί και σε ό,τι αυτό το βαθμό εναρμόνισης υπάρχει μια συμβαστική πρόταση. Πώς να το πω, προτείνεται μια ελάχιστη εναρμόνιση ως αρχή. Αλλά με πολλές εξαιρέσεις τελικά όπου τελικά ορίζεται πού υπάρχει πλήρης εναρμόνιση. Αυτός είναι ο συμβιβασμός ώστε να είναι ικανοποιημένοι και αυτοί που θέλουν την πλήρη εναρμόνιση και αυτοί που θέλουν την συμβιβασμό, εναρμόνιση. Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι υπήρχε ένας πολιτικός στόχος κοινός σε όλους. Το υφιστάμενο δίκαιο να μην υποβαθμιστεί κανένα κράτος μέλος. Αυτό ήταν το πρόβλημα με την πλήρη εναρμόνιση. Δεν μπορεί κανείς να περιμένει ότι θα υπήρχε πλειοψηφία ούτε στο Συμβούλιο, όπως και δεν θα υπήρχε στο Κοινοβούλιο ε, η εναρμόνιση προς τα πάνω, ε, στο το ανώτερο επίπεδο, αλλά εναρμόνιση σε ένα υψηλό επίπεδο ε, δεν ήμουν ε, παρούσα στις τελευταίες διαπραγματεύσεις, αλλά κατάλαβα καλά, αύριο θα αποφασίσουμε τα εξή δύο. Σε μια σειρά, ε, για μια σειρά δικαιωμάτων, τα κράτη-μέλη που έχουν ε, για αυτά τα κρυφά ελαττώματα, παραδείγματος χάρη ένα δικαίωμα ή μια διάταξη, τη διατηρούν μέχρι το σημείο που θα τεθεί σε ισχύ η οδηγία. Και υπάρχει μια δεύτερη, και τα λέω για περίπλοκα γιατί είναι περίπλοκα τα πράγματα, υπάρχει δεύτερη εναλλακτική, νομίζω για τις προθεσμίες ήταν ε, για τις ψυχικές περιπτώσεις, που δεν θυμάμαι ακριβώς, Εδώ επιλέγουμε την ελάχιστη δυνατή εναρμόνιση. Έχουμε τα έξι χρόνια, μια προθεσμία Αφήνουμε δηλαδή την ελευθερία στα κράτη-μέλη αν θέλουν να έχουν αυτά τα 6 χρόνια ή όχι. Αυτή ε, ήταν ε, η συμβαστική πρόταση ε, στους συναδέλφους ΙΜΚΟ χθε. Τώρα για το Συμβούλιο δεν ξέρω πώς θα έρθει το διέξοδο γιατί έχουμε μία διπλή μειοψηφία που μπλοκάρει και για την πλήρη και για την ελάχιστη εναρμόνιση ε, και εκεί το πρόβλημα. Και δεν βλέπω, ε, γιατί δεν υπάρχει καμιά κοινή θέση από το Συμβούλιο ακόμη, δεν βλέπω πότε θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι σε αυτό τον τομέα. Και αυτό συνδέεται με αυτό που έλεγα πάντοτε. Δεν μπορούμε να αφήσουμε για τα ενσώματα αγαθά ή τα σώματα μέσα ένα μέρος των ψηφιακών, ε, του ψηφιακού περιεχομένου. γιατί θα πληγεί η εσωτερική αγορά αν ισχύουν διαφορετικοί κανόνες ε, για διαφορετικά τμήματα του ψηφιακού περιεχομένου των ψηφιακών προϊόντων. και επίσης επειδή δεν υπάρχει ε, μια ενιαία νομοθεσία να έχουμε τελείως διαφορετική νομοθεσία στο κάθε κράτος μέλος και αυτό βλάπτει. Ε, αυτά είναι πολύ πλοκά, είναι πάντως και συναρπαστικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες αυτές. Θα περιμένουμε αναγωνίως να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό στην πράξη Νομίζω όμως ότι οι δικηγόροι είναι ήδη έτοιμοι γι' αυτό. Τελειώσαμε λοιπόν το 10, το 11 το έχουμε τελειώσει. Το 10 είναι απλώς ε, ενημερωτικό. Οπότε εδώ ολοκληρώνεται το δημόσιο κομμάτι της ε, συνεδρίασής μας σήμερα. Θα συνεχίσουμε και κλειμένων των θυρών με δύο σχετικά σύντομα σημεία, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα φύγουν ε, οι συνάδελφοι. Πρέπει να είμαστε τουλάχιστον 8, οπότε δεν πρέπει να φύγετε. Είμαστε 9 αυτή τη στιγμή, επειδή ε, θα ψηφίσουμε. Οπότε, αν μπορείτε παρακαλώ να καθίσετε για μερικά ακόμη λεπτά, θα είναι πολύ ευγενικό εκ μέρου σας. Κλείνουμε λοιπόν το δημόσιο τμήμα των εργασιών μας. Παρακαλώ όσους δεν δικαιούνται να βρίσκονται ε, στην κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση να αποχωρήσουν.